Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας ε, διάταξης. Προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε σχέση με την ανανέωση του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Το λόγο έχει η συντάκτρια η κυρία Μακέιβον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε Στυλιανίδη, από το Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Βρισκόμαστε στη βραδινή βάρδια, αλλά ωστόσο πρέπει να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ξέρω πως συμφωνείτε όλοι. Θέλαμε η συζήτηση αυτή να λάβει χώρα σήμερα, διότι θέλαμε να δούμε μια πραγματική δέσμευση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη για να γίνουν αλλαγές σχετικά με την χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα. Θέλουμε να ληφθεί στα σοβαρά η ε, ατζέντα για την ισότητα και όχι απλά να μένουν στα λόγια τα θεσμικά όργανα. Θέλουμε να δούμε αυτή την ε, αλλαγή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το τελευταίο πρόγραμμα ε, ανακοίνωσε πως τα αποτελέσματα ήταν αποσπασματικά και δεν είχαν αρκετά στοιχεία και πως βασίστηκε στην θέληση λίγων μόνο ε, προσώπων παρά σε μια συλλογική ανταπόκριση. Θέλουμε λοιπόν να δούμε την αλλαγή. Πολύ φοβάμαι όμως πως θα αρχίσω τα σχόλιά μου με αρνητική ε, χρειά. Θα ήθελα ε, να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να δημοσίευσει μια ανακοίνωση για το νέο σχέδιο δράσης έτσι ώστε να δώσει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό στίγμα. Ένα μήνυμα ότι η ισότητα έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντική και ότι η χειραφέτηση των γυναικών πρέπει να μπει πιο ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ζητήσαμε ε, περισσότερη επικοινωνία, διότι ακούσαμε πολλές φήμες οι οποίες δυστυχώς αληθεύουν ότι αυτό που πρόκειται να δημοσιεύσει η Κομισιόν είναι ένα έγγραφο εργασίας και όχι μία ανακοίνωση όπως προβλεπόταν. Και πράγματι μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο εργασίας για το θεματολόγιο της ισότητας. Μίλησα με πολλούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άκουσα τα επιχειρήματά τους, δεν επιθυμούν να ε, δημοσιεύουν μία ανακοίνωση μετά την άλλη, αλλά πιστεύω πως ε, αυτή η συζήτηση για το τι έγγραφο θα είναι μας εμποδίζει, μας καθυστερεί. Ας μιλήσουμε καλύτερα για την αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος, διότι εδώ πιστεύω πως θα δείτε ότι πρέπει να ληφθεί στα σοβαρά αυτό το έγγραφο. Η αξιολόγηση λέει ότι τα κίνητρα ε, για να ε, γίνει μια αρχή, ε, είτε από τις Βρυξέλλες είτε από τις αντιπροσωπείες, έλειπαν. Δεν υπήρχε θέληση. Δεν υπήρχαν κίνητρα αποτύχαμε από το να κάνουμε κάτι. Εάν είχε δημοσιευθεί μια ανακοίνωση θα είχε εγκριθεί από όλο το σώμα των επιτρόπων και αυτό που χρειάζεται είναι εμείς να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όμως δυστυχώς αυτό είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ανακοίνωση και όχι ένα έγγραφο εργασίας. Χρειάζεται λοιπόν ένα σχέδιο δράσης. Όμως με τον τρόπο που έγινε δεν ήταν και ο πιο σωστός τρόπο για να αρχίσει μια συζήτηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να περιληφθούν ε, τα θέματα Ευρωπα... στο έργο της Επιτροπής. Ξέρω πως ο Επίτροπος είναι φεμινιστής, είναι δεσμευμένος να το κάνει αυτό. Ξέρω ε, πως ε, και η Προεδρία του Συμβουλίου έχει δεσμευτεί να προχωρήσει το θέμα της ισότητας. Γι' αυτό, λοιπόν, σύμφωνα με το ψήφισμά μας, αυτό που ζητούμε είναι συγκεκριμένε πολιτικές, συγκεκριμένη οικονομική πόρη, ισότητα, η ισότητα να μπει στην ατζέντα των αντιπροσωπιών, να δοθεί περισσότερη έμφαση στις αξιολογήσει, να συμπεριληφθεί στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις τρίτες χώρε, να συμπεριληφθεί στον, στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό, να ε, σταματήσουν οι διακρίσει στους μισθούς και στην οικονομική και επαγγελματική ζωή. Να υπάρχει ίση πρόσβαση στην υγεία, ίση πρόσβαση στα ε, σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Κύριε Επίτροπε, αυτό που θέλω να ακούσω από εσάς είναι πώς θα τεθούν σε ισχύ αυτά τα σχέδια και τη ε, χρηματοδότηση. Τι θα γίνει με την παρακολούθηση των εδράσεων και τέλος θα ήθελα αυτή η συζήτηση να γίνει στο ευρύτερο πλαίσιο των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Πριν από δύο εβδομάδες στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκαν αυτοί οι στόχοι. Ο στόχος 5 μάλιστα αναφέρει την ισότητα και την χειραφέτηση των γυναικών. Αυτοί οι στόχοι πρέπει όμως να μεταφραστούν σε δράσεις εδώ. Πολλοί λένε πως χρειάζονται δείκτες να το, για να γίνει αυτό. Πολλοί λένε επίσης ότι χρειάζεται να γίνει μια επανάσταση να συμπεριληφθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια. Όμως χρειάζεται πληροφόρηση, διότι αν δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χρειάζεται να συμπεριληφθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια, χρειάζεται να νιώσουν αυτήν την αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να αφήσουμε ένα έργο πίσω μας και έχετε την πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να το πράξετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Συγήτρια. Ο κύριος Νικολάς Σμιτ από το Συμβούλιο. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία μου, θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Κι εγώ είμαι φεμινιστής, γιατί ασχολήθηκα στην προηγούμενη μου ζωή με την ε, συνεργασία για την ανάπτυξη και είμαι πεπισμένος ότι η ανάπτυξη περνάει από τις γυναίκες και από την εκπαίδευση των γυναικών και από την ε, συμμετοχή των γυναικών στον οικονομικό ιστό. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών εντάσσεται στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη προστατεύουν και προωθούν τα δικαιώματα της γυναίκας και αυτό και στις εξωτερικές δράσεις. Το 2015 είναι σημαντική χρονιά γιατί εγκρίθηκε το αναπτυξιακό πρόγραμμα του 2015 αλλά και το, τη 15η επέτειο του ψηφίσματος 1325 των Ηνωμένων Εθνών και της ε, δήλωσης και του προγράμματος δράσης υπέρ των γυναικών. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους σε ένα θέμα ύψης της σημασίας. Κατά το δεύτερο εξάμεινο η Λουξεμβουριακή Προεδρία προωθεί τις εργασίες στο Συμβούλιο για την ισότητα των φύλων και την ανάπτυξη βασίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα πλαίσια της ε, ανάπτυξης. Αυτή θα είναι και η προτεραιότητά μας και στα κράτη-μέλη και στην εξωτερική μας πολιτική. Στο Συμβούλιο συνεργαζόμαστε δραστήρια με τα κράτη-μέλη και με την ΕΙΕΔ για να υποβάλουμε ένα νέο πρόγραμμα δράσης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την χειραφέτηση των γυναικών. Παγκόσμια έχουν γίνει, έχει γίνει πρόοδος για την ισότητα των δύο φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών και των ε, νέων κοριτσιών. Τα νέα κορίτσια συμμετέχουν ε, στην εκπαίδευση και στην οικονομική ζωή. Όλο ένα και περισσότερες ε, γυναίκες έχουν πρόσβαση στην υγεία και η ε, θνησιμότητα κατά τη γέννηση έχει μειωθεί. Όμως η πρόοδος δεν είναι τόσο γρήγορη όσο θα θέλαμε και είναι άνηση ανάλογα με τις περιφέρειες της χώρες αλλά και μέσα στην ίδια χώρα. Κάθε χρόνο παντού στον κόσμο δυστυχώς καταπατούνται τα δικαιώματα των γυναικών και των ε, νέων κοριτσιών. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, διακρίσεις ε, ούτε σεξουαλική εκμετάλλευση δεν πρέπει να υπάρχει γενετικό, γενετικός ε, παρέμβαση στις ε, γενετικές προτιμήσεις, ούτε ακροτηριασμός γενετικών οργάνων. Γι' αυτό θα θέλαμε το νέο πρόγραμμα δράσης, το οποίο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να είναι ένα ουσιαστικό μέσο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών και των νέων κοριτσιών που είναι θύματα διάκρισης θεωρούμε ότι το νέο πρόγραμμα δράσης είναι υποχρεωτικό μέσα στα πλαίσια συνεργασίας των κοινοτικών φορέων. Χρειάζεται ε, να λάβουμε υπόψη το institutional cultural shift και επιτόπου δηλαδή να εντάξουμε και τα δύο φύλλα εγκάρσια σε όλους τους τομείς. Τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο Συμβούλιο επί θέματος. Το θέμα της ισότητας των δύο φύλων και της ανάπτυξης θα μας απασχολήσει μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών στις 26 Οκτωβρίου. Άρα θα προωθήσουμε και το νέο πρόγραμμα δράσης ισότητας των δύο φύλων. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν μάχη για την ισότητα των δύο φύλων και η Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Στυλιανίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Εδώ έρχομαι να σας μιλήσω εκ μέρους του συνεργατικού συνοδέλφου, θα ελπίζω κύριε Μακάβα να μπορέσω να σας ε, καλύψω γιατί προσπάθησα να σας ε, εξηγήσω ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί αυτή η η καθυστέρηση που έχουμε όσον αφορά το να πετύχουμε την ισότητα ε, έρχεται σε με το ότι εμείς θέλουμε να έχουμε κάποιες δράσεις που να έχουν επιπτώσεις, κάποια μέτρα με χρηματοδότηση, με εμπειρογνωμοσύνη αλλά επίσης και με βούληση πολιτική για κάθε πολιτική αλλά και όσον αφορά την ε, εξωτερική δράση και αναπτυξιακή πολιτική αυτό θεωρούμε ότι υλοποιείται τώρα που έχουμε ε, τις νέους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο η υπηρεσία ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε κατά νου καινούργια υπηρεσία της Δράκης όταν, όταν εγκρίναμε αυτό το καινούργιο πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών μέσω των όσων θα γίνουν στην περίοδο 16 έως 2020. Αυτό λάβετε υπόψη και δείτε στην ουσία αυτών των προτάσεων ότι πρόκειται για κάτι το φιλόδοξο, για κάτι το οποίο διαδέχεται το σημερινό πρόγραμμα δράσης ε, γιατί σύντομα αυτό πρόκειται να εκπνεύσει. Οπότε τώρα έχουμε κάποια φιλοδοξία που μπορείτε να διαπιστώσετε στο θεματολόγιο και στο τι καλύπτουμε γεωγραφικά. Θα ισχύσει αυτό το καινούργιο ε, πρόγραμμα για όλες τις εξωτερικές πολιτικές μας και για την εμπορική πολιτική και για την ανθρωπιστική αρρωγή. Επίσης όλα αυτά θα ισχύσουν και για όλες τις ε, χώρες εταίρους μας αλλά και για κάποιες ε, δύσκολες καταστάσεις, ή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκες και θα δούμε επίσης τι γίνεται για εκεί που υπάρχει μετασχηματισμός του, του σε γυναίκα, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε κάθε δυσμένη διάκριση, κάθε βία και έτσι αυτές οι κοπέλες να έχουν ισότητα προσβασιμότητας σε όλες τις ε, οικονομικές διαδικασίες, τους πόρους και να έχουν έτσι χειραφέτηση κοινωνική και πολιτική. Σας τονίζω το εξή. το επίπεδο φιλοδοξίας μας, το επίπεδο αυτού του νέου ε, πλαισίου δεν έχει θυγεί από τα όσα διαπιστώνονται στο έγγραφο εργασίας. Έχουμε κάνει μια αλλαγή που θεωρούμε ένα θετικό βήμα και έτσι θεωρούμε ότι οι υπηρεσίε τη Επιτροπή και τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα συνεργαστούν. Θα συνεργαστούν με αποτελεσματικότητα, με συνέπεια και στρατηγικά. Και έτσι ε, τα δικαιώματα των ανηλίκων γυναικών και ενηλίκων γυναικών πρόκειται να κατοχυρωθούν και γι' αυτό θέλουμε και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν αυτή μας την προσέγγιση μέσω των αντιστοίχων αποφάσεων που θα λάβει το Συμβούλιο και όλα αυτά να είναι εφαρμόσιμα και να αποτελέσουν μια συντονισμένη προσπάθεια σε ενωσιακό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκείνο να συμπαρασταθεί σε αυτή την συλλογική προσπάθεια και έτσι να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα καταφέρουμε να αποσπάσουμε και για αυτό και είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει από το περιβόλι μας να αρχίσει η αλλαγή. Θα, δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει το πνεύμα που επικρατεί στα θεσμικά όργανα και αυτό να γίνει με κάποιο είδους αντίστοιχη ε, διακυβέρνηση για όλα τα θεσμικά όργανα, για όλα τα ε, ε, κράτη-μέλη και έτσι να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά το στόχο μας για την ισότητα των φίλων. Θα θέλω να είστε βέβαιοι ότι ό,τι έχει ξεπεραστεί ε, θα πρόκειται ε, να αντικατασταθεί από συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη εις ε, την υπηρεσία μας, της αντιπροσωπείες της Ένωσης στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υπάρξει και στόχοθετημένη κατάρτιση αυτού του προσωπικού. Επίσης υπολογίζουμε ποσικά τους στόχους και γι' αυτό και έχουμε πει ότι θα διαθέσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ για τα σχετικά μέτρα, ούτως ώστε να πετύχουμε την ισότητα των φύλων. Και ακόμα περισσότερα θα εκταμιευθούν μέσω κάποιων προγραμμάτων που θα αντιμετωπίζουν ε, διάφορους άλλους τομείς και άλλες προτεραιότητές μας σε γεωργία, ενέργεια, ε, δικαιοσύνη, μετανάστευση. Όμως, εμείς σε όλες αυτές τις πολιτικές πρόκειται να λαμβάνουμε υπόψη αυτή την πολιτική για τα δικαιώματα γυναικών και ανηλίκων γυναικών επίσης. Ε, θα υπάρξει κάποια ε, δομή για κοινοποίηση αποτελεσμάτων, οπότε όλοι σε όλα τα επίπεδα να λογοδοτούν για το τι πετυχαίνουν γιατί δεν πετυχαίνουν. Οπότε, εν κατακλείδη, θέλω να σας επαναλάβω ότι εμείς είμαστε δεσμευμένοι 100% ώστε να έχουμε πλήρη υλοποίηση αυτού του καινούργιου πλαισίου πολιτικής για τα δύο φύλλα και θα υλοποιήσουμε όλες αυτές τις σκοπόμενες αλλαγές και ελπίζουμε ότι θα έχουμε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια το Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο πρόκειται να μας βοηθήσει σε αυτή την πρωτοβουλία της Επιτροπής. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed, Mr. Commissioner. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Αρχίζουμε τώρα με τους εκπρόσωπους των πολιτικών ομάδων και αρχίζουμε εκ μέρου του ΕΛΚ ο Ντάβορ Ιβο Στίερ. Έχετε μισή λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, ε, την εισηγήτρια, να την συγχαρώ και να συγχαρώ επίσης και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο σχέδιο δράσης, έτσι όπως το ψηφίσαμε στην Επιτροπή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχέδιο αυτό και πιστεύω πως αξίζει πραγματικά να έχουμε μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε, 14 εκατομμύρια κορίτσια παντρεύονται καταναγκαστικά, 22 εκατομμύρια κορίτσια δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες ε, στερούν από τις γυναίκες πολιτικά δικαιώματα, επαγγελματικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα. Υπάρχουν κορίτσια τα οποία βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μόνο και μόνο για το φίλο τους. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει τον κόπο για πάρα πολλούς λόγους να επενδύσουμε στις γυναίκες. Οι γυναίκες δίνουν το 90% του εισοδήματός τους πίσω στην οικογένεια και όμως κερδίζουν το 40% ε, σε ορισμένες χώρες ε, από τους ε, άνδρες στην ίδια θέση. Χρειάζεται λοιπόν να πούμε σαφώς ότι χρειάζεται δράση και ότι αξίζει να ενισχύσουμε τον ρόλο και την θέση των γυναικών. Γι' αυτό και το 2014 στο ψήφισμά μας τονίσαμε σαφέστατα πως οι γυναίκες παίζουν έναν κεντρικότατο ρόλο στην νέα πολιτική ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, ο Ντόρου Κλάουδιαν Φρουντζούλιτσα. Έχετε τρία λεπτά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεδομένης της σημασίας της χειραφέτησης των γυναικών, όχι μόνο ως ε, δεδομένο ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και ως μέρος της, ε, των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης πιστεύω πως η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 για το μέσο αναπτυξιακής συνεργασία είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ε, αξιολογήσουμε τα προγράμματα για τις γυναίκες και τα κορίτσια και να γίνουν οι αναγκαίες αναπροσαρμογές ε, του προπολογισμού. Οι στόχοι της χιλιετίας ε, τονίζουν την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών και της ισότητας των φίλων της ε, υγείας των γυναικών. Δυστυχώς όμως πολλοί από αυτούς απέχουν ε, πολλοί από το να επιτευχθούν. Η πρόοδος είναι αργή και δεν έχει γίνει με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Η εφαρμογή του προγράμματος από το 2010 μέχρι το 2015 δείχνει πως χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα χειραφέτησης των γυναικών και χρειάζεται ανανέωση της δέσμευσης και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από τα λαθεσμικά όργανα για να βελτιωθούν, βελτιωθούν οι προδιαγραφές για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Επίσης χρειάζεται να δοθεί περισσότερη σημασία στους οργανισμούς ε, των γυναικών και να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών. Πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε οι γυναίκες να ε, αποκτήσουν ισότητα επαγγελματική σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους και να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να αποτραπούν οι διακρίσεις κατά των γυναικών βασισμένες στην ε, μητρότητα ή στο, στην ε, κατάσταση ε, στη συζυγική τους κατάσταση. Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναπτυξιακή συνεργασία, η ανθρωπιστική βοήθεια, το εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το μεταναστευτικό ζήτημα, το άσυλο και ε, πολλές άλλες πολιτικές ε, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις γυναίκες. Πρέπει επίσης να να πηγαίνουν πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να ενισχυθεί η σωστή, η χρηστή διακυβέρνηση και να καταπολεμηθεί ε, ο βιασμός των γυναικών ως ε, όπλο αποσιώπησης της φωνής τους. Πρέπει να φροντίσουμε οι ένοχοι να βρεθούν υπόλογοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Και μόνο όταν αντιμετωπίσουμε επιτυχώς όλα αυτά τα προβλήματα μόνο όταν επανέλθουν οι ανθρώπινες αξίες εκεί που πρέπει να βρίσκονται, μόνο τότε θα έχουμε μια δίκαιη και ίση κοινωνία για όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχει το λόγο τώρα εκπρόσωπος ε, της ομάδας ECR, ο κύριος ε, Μπρανισλαβ Σκρίπετ. Έχετε ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ Σωστό τόπους η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τις, χώρες, ε, τις τρίτες χώρες. Όμως η βοήθεια αυτή θα επιβάλλει ιδεολογίες ε, σχετικά με το φύλλο που διαφέρουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε πως ε, ο πληθυσμός των φτωχότερων χωρών, των χωρών του τρίτου κόσμου, χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη ελευθερία, περισσότερη δικαιοσύνη περισσότερο αυτό παρά καταπολέμηση των στερεοτύπων. Χρειάζεται να σεβαστούμε τα ήθη και τα έθιμα των ε, τρίτων χωρών και όχι να τους επιβάλλουμε τις δικές μας ιδεολογίες και τα δικά μας πρότυπα και τρόπο ζωής. οι διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να επασχίσουν για την ε, πλήρη ένταξη όλων των κοινωνικών στρωμάτων, ανδρών και γυναικών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ε, διεθνείς θεσμοί να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπαστερετσέα Μπεατρίθ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Σμιτ, και στη Λιανίδη. Κυρία Μακ Έιβαν, σας ευχαριστώ πολύ. Έχει μεγάλη σημασία η ισότητα των δύο φίλων. Πρόκειται για το στόχο υπαριθμών 5. Οι γυναίκες είναι το ίμιση και κάτι παραπάνω του πληθυσμού στον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για ε, πλειοψηφία Πρόκειται για βασικό ανθρώπινο δικαίωμα η ισότητα, έτσι ώστε να ευημερίσουν και οι γυναίκες. Οι 193 χώρες που έχουν προσυπογράψει τάσσονται υπέρ αυτών των στόχων. Θα πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο για τους στόχους που ορίσαμε εδώ και δύο εβδομάδες θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών. Μία στις τρεις γυναίκες και στην Ευρώπη υφίσταται σεξουαλική ή ψυχολογική βία. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη βελτίωση της κατάστασης των ε, γυναικών μέσα στα πλαίσια της Σύμβασης της Ισταμπούλ. Έχει μεγάλη σημασία όμως η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση είναι ύψης της σημασίας διότι τα νέα κορίτσια, τα κορίτσια θα μπορέσουν να συμμετάσχουν αργότερα στην παγκόσμια ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρξει ένα παγκόσμιο ταμείο για την εκπαίδευση μέσα στα πλαίσια του στόχου υπαρθμών 4 η πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσα στα πλαίσια της ισότητας των δύο φύλων. Όπως είπε ο ειδικό ε, ε, εμπειρογνώμων των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει ίση πρόσβαση, γιατί μόνο αν συμμετέχουν τα κορίτσια θα περάσει το μήνυμά τους. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, η κυρία Σάντσες Καλντεντέ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ισότητα των δύο φύλων είναι βασικό, θεμελιώδες δικαίωμα. Όμως η μισθή των γυναικών είναι 30% κατώτερη από των ανδρών και μία από τις ε, τρεις γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική ή ψυχολογική βία και δεν έχει πρόσβαση στην εργασία. Δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Το πρώτο πρόγραμμα δράσης δείχνει μεγάλες ελλείψεις. Η έκθεση που θα ψηφίσουμε αύριο είναι ιδιαίτερα ε, φιλόδοξη και θα την υποστηρίξουμε. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ενίσχυση των γυναικών σε όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν προσκόμματα ε, ε, σε πρόσβαση σε οποιαδήποτε, οποιοδήποτε ομέα. Δεν θα πρέπει η γυναίκα να θεωρείται εξόριστη παντού. Εμείς πραγματικά είμαστε θύματα. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στην δωρεάν άμβλωση. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει ισότητα. Επίσης θα πρέπει να υποστηριχτεί αυτό το σχέδιο από το Διευθυντήριο των Επιτρόπων. Διαφορετικά θα είμαστε πάντα πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ευχαριστώ πολύ. Εξ των Πρασίνων, ο κύριος Σεμπαστιά Ζόρντι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ θλιβερό να βλέπουμε την αίθουσα τόσο άδεια. Ποτέ δεν την είχα δει τόσο άδεια. Αυτό συμβαίνει με το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, αλλά αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξαλείψουμε τις ε, διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες παγκοσμίω. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο μία δήλωση προθέσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι αυτό το έγγραφο είναι έγγραφο εργασίας, δεν είναι μία ανακοίνωση της Κομισιόν και δεν μιλάμε για αύξηση των πόρων για την ισότητα των δύο φύλων έτσι μιλάμε και παραμένουμε στα λόγια. Θα εγκρίνουμε το κείμενο, αλλά θέλουμε περισσότερα κονδύλια και περισσότερες γραμμές του προϋπολογισμού. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική να προωθήσει αυτό το θέμα σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Από την ομάδα ΙΕΝΕΦ η κυρία Τροσκίνσκι για δυόμιση λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Μα και πάλι μία έκθεση γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει ένα ιδεολόγημα. Τη βία κατά των γυναικών αλλά στο πρόγραμμα δράση 2010-2015 δεν, ε, ε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την φυσική και ψυχολογική ακαιρεότητα των γυναικών. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι αιστείες βίας ιδιαίτερα στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο ιδιαίτερα στις χώρες του Ισλαμικού φονταμενταλισμού επιβάλλεται η βία. Ο ημάμις της Μπρέστ μίλησε στη Γαλλία σε διάφορες εφημερίδες εάν η γυναίκα βγαίνει χωρίς τη μαντίλα, τότε δίνει το δικαίωμα στους άνδρες να ε, καταχραστούν της καλοσύνης της. Τι μπορούμε να πούμε για τις χώρες όπου πολλούνται οι γυναίκες, αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίου. Δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για την Boko Haram ή το Ισλαμικό κράτος που δεν δέχονται τα δικαιώματα των γυναικών. Πρόκειται για τρομοκρατικές οργανώσεις που δρούν οπουδήποτε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι χώρες του Περσικού κόλπου ε, προβάλλουν αυτή τη στάση στην ε, Αγία Πετρούπολη 700 γυναίκες από ολόκληρο τον κόσμο σε, από ΜΚΟ, πανεπιστήμια και ούτω καθεξής ε, δώσαν μαρτυρία για το τι συμβαίνει σε προσωπικό, τι υφίστανται σε προσωπικό ή και επαγγελματικό επίπεδο. Μίλησαν για βιαιότητες, για βιασμό και για ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων. Οι γυναίκες θα θέλαν να τις βοηθήσουμε στη χώρα τους ή να βοηθήσουμε την κυβέρνησή τους να ε, καταπολεμήσει την τρομοκρατία ζητούμε ειδική δράση για να ενισχύσουμε τα ε, δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Οι αναπτυσσόμενες χώρες το χρειάζονται αυτό. Και μέχρι πού θα κινηθείτε μέσα στα πλαίσια του άκρα του ιμπεριαλισμού σας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκέρλινγκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ 100% όσον αφορά αυτή τη δράση για την γραφεία των γυναικών και αυτό το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φίλων της ε, Ένωσης. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αναδειχθεί η σημασία αυτού της υπόθεσης, ε, αυτό που είπε η κυρία Μακάβαν, για αυτό να εγγύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τώρα το ECR και οι τόρε. Θέλουμε να είναι η γυναίκα στο επίκεντρο των διεθνών ε, εξελίξεων για την ανάπτυξη και πιστεύουμε ότι έτσι υπάρχει θετική επίδραση όσον αφορά την κατανόηση της φτώχειας, την ανάπτυξη και ότι έτσι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Επίσης, είναι πάρα πολύ θετικό ότι το πρόγραμμα τώρα έχει καινούργια όθηση, ανανεώνεται, αλλά τα προβλήματά μας είναι ότι δεν έχουμε αρκετή έμφαση στην πληροφόρηση και την μεθοδολογία και θα προτιμούσαμε να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες και να δίνουμε περισσότερα χρήματα όσον αφορά ε, κυριολεκτικά τις ε, δράσεις. Επίσης ε, εστιάζεται περισσότερο ε, στην λάθος προσέγγιση ε, αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι καλύτερη βρετανική προσέγγιση όσον αφορά την πολυμερή αναθεώρηση της ε, βοήθειας γιατί είναι το πιο σημαντικό θέμα αυτό. Ο πρώτος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Κάθριν Μπίρντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ Λίντα Μάκαβαν για τα όσα έκανες, γιατί ήδη θεωρούμε ότι η ισότητα σημαίνει και ισότητα των φίλων. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό αυτό να είναι βασικό στις στρατηγικές μας και ιδίως φέτος που έχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει η γυναίκα να μην ε, έχει τον, τον, ε, την απειλή της βίας και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες. Έχουμε συγκρούσεις, έχουμε στην ε, Νιγηρία, την Μπόκα Χάραμ εκεί, έχουμε ε, βιασμού στη Συρία επίσης. Τι βλέπετε οι γυναίκες εκεί φεύγουν τόσο από τον πόλεμο και λοιπά και πολλά άλλα. Αλλά είδαμε τι γίνεται, ότι από αυτή τη βία έχουμε πάρα πολλές εγκυμοσύνες και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μα λέει ότι το, έχουμε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των δικαιωμάτων που θα πρέπει να επιτρέψουν την ελεύθερη άμβλωση. Και αν μην συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, θα πρέπει οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε προστασία, σε υποστήριξη και να μπορούν να έχουν δικαιώματα αναπαραγωγικά και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό όσον αφορά την ελευθερία τους και τη χειραφέτησή τους. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν αναπαραγωγικά δικαιώματα και να έχουν όταν χρειάζεται κάποια ασφαλή και νόμιμη αμβλώση. Είναι βασικό αυτό, να υποστηρίξουμε τις γυναίκες στις περιοχές των πολέμων και για εκείνες οι οποίες φεύγουν να γλιτώσουν από την βία. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε και τώρα για την ε, γκουα. Κύριε Φορέντζα, το λόγο. Έχετε ένα λεπτό, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και δυνάμει αυτών των συνθήκων και των στρατηγικών που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 που ο ΙΕ δημοσιοποίησε ε, πρόσφατα νομίζω θα πρέπει το κοινοβούλιο μας να διαθέσει τους πόρους που υπάρχουν και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει το δεύτερο στόχο και στο επίπεδο της Ένωσης αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών να έχουμε ε, αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη και έτσι να μπορούμε να βοηθήσουμε και σε επίπεδο ε, υγεία, σε επίπεδο υπηρεσιών ε, βιώσιμη ανάπτυξη ούτως ώστε να μπορούν οι γυναίκες να διαλέξουν τι θα κάνουν και να έχουν ίση ίσα δικαιώματα στη δουλειά με τους άντρες συναδέλφου και οπότε ε, ε, έτσι να πετύχουμε την ισότητα των γυναικών και να δούμε ε, το ότι αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ κατεπήγον. Επίσης προτείνω όλα τα κράτη-μέλη, κυρίως της Νότιας Ευρώπης, να φτιάξουν αυτό τον δίκτυο, αυτό το κριτήριο της ισότητας και αυτό να χρησιμοποιηθεί και σε περιφερειακό επίπεδο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πολιτική αποτελεσματική και επίση στα πλαίσια αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη να έχουμε μια ανάπτυξη και αυτό να ισχύσει και στι αναπτυσσόμενε και στι αναπτυγμένε χώρε. Όλα αυτά μα αφορούν άμεσα. Ο Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα αρχίζει η διαδικασία του Catch the Eye. Έχουμε δύο μια κυρία πρώτα. Όχι, όχι, λέει ο πρόεδρος. Είναι ο κύριος Ρικάρντο Σάντος. Το πρόγραμμα δράσης 10-15 ε, μας οδήγησε σε μια νέα πολιτική αναπτυξιακού χαρακτήρα. Όμως θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να έχουμε νέα προσέγγιση, νέες προσεγγίσεις. Το πρόγραμμα 15-20 θα πρέπει να είναι φιλόδοξο και συνεκτικό. Θα πρέπει να ε, συλλέξουμε τους ε, κοινωνικούς ε, στόχους και να τους εντάξουμε να προωθήσουμε την ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε ε, αυτές τις δραστηριότητες και μέσα στο, στις εμπορικές μας ε, συναλλαγές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταπολεμήσει τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα που παρατηρούνται στους χώρους δουλειάς, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη χειραφέτηση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην περίοδο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης που διανύουμε παρατηρούνται έντονες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών καθώς και διαφορές σε μισθούς και συντάξεις ανάμεσα στα δύο φύλλα σε όλο τον κόσμο επιπλέον τα επίπεδα ανεργίας των γυναικών ξεπερνούν κατά πολύ αυτά των ανδρών γεγονός που δείχνει ακόμη πιο έντονα τις διακρίσεις όσον αφορά τα κριτήρια πρόσληψης των εργαζομένων. στη φτωχοποιημένη από το μνημόνιο ελλάδα οι γυναίκες είναι τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης. έτσι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στο πρώτο τρίμηνο του δύο είναι τριάντα έξι έναντι είκοσι πέντε των ανδρών τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης οφείλουν να παλέψουν προκειμένου να εξαλειφθούν οι μισθολογικές διαφορές στον αναπτυσσόμενο κόσμο να επιβάλλουν τη διαφάνεια στα σύνταξιοδοτικά συστήματα όσον αφορά τα δύο φύλλα. επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών σε σχέση με την μητρότητα και να αντιταχθούν στην άδικη απόλυση γυναικών εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αναπληρωτής Μαριάς. now Ήρθε η ώρα λοιπόν για τον προσκεκλημένο μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε Στυλιανίδη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ την συνάδελφο Λίντα Μακάβαν για την αφοσίωσή της σε ένα τόσο απαιτητικό ζήτημα με τόσες μεγάλες προκλήσεις. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ ειλικρινά για αυτή την ε, πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων σε αυτούς τους ε, δύσκολους καιρούς. Αυτό δείχνει πως ε, οι θέσεις μας βρίσκονται πάρα πολύ κοντά η μία στην άλλη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την βελτίωση της ζωής των γυναικών και των κοριτσιών στις ε, χώρες εταίρους μας. Ελπίζω οι ανησυχίες σας ε, να ε, αντικατοπτρίζονται στο νέο πλαίσιο δράσης μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το διάλογό μας και την εφαρμογή του. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι έχετε δείξει μια γενικότερη μεγάλη αφοσίωση στα ζητήματα των γυναικών, ιδιαίτερα μάλιστα φέτος που γιορτάζουμε την 20η επέτειο της πλατφόρμας του Πεκίνου και την 50η επέτειο του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Κάτι το οποίο θα εγκριθεί στα πλαίσια της, ε, του θεματολογίου για την αβιώσιμη ανάπτυξη του 2030. Δεν πρέπει κανείς να μείνει πίσω, ιδιαίτερα οι γυναίκες και τα κορίτσια. Το θεματολόγιο του 2030 είναι ένα οικουμενικό πλαίσιο που έχει πολύ φιλόδοξους στόχους και επίσης επιβεβαιώνει εκ νέου το ρόλο της χειραφέτησης των γυναικών. Οι γυναίκες που είναι κλειδί και πρωτοπόροι στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης πριν από δύο εβδομάδες στη Νέα Υόρκη τόνισε πως αυτό που επιθυμούμε είναι να ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών γίνονται σεβαστά πανταχώθεν και όπου ο καθένας έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στο έπακρο των δυνατοτήτων του στην κοινωνία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι δεσμευμένη 100% για να πραγματοποιήσει αυτήν την υπόσχεση μέσω αποτελεσματικής εφαρμογής ε, του ε, πλαισίου για τα δύο φύλλα και με τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών, της κοινωνίας των πολιτών, των ε, διεθνών και μη κυβερνητικών οργανισμών, των επιχειρήσεων και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Και φυσικά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηριζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γίνει ο πιο σημαντικός εταίρος μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο για να ολοκληρώσω.